σας. Είμαστε υπέρ της πρόθεσης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Μάλιστα κάτι τέτοιο περιλαμβάνεται και στο σχέδιο δράσης μας, γιατί έχουμε σχέδιο δράσης για ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία που πλησιάζει στο τέλος του. Τώρα εξετάζουμε το νέο σχέδιο δράσης που θα καλύπτει την περίοδο 2015-2019. Και τους τελευταίους μήνες ακριβώς ασχοληθήκαμε με την ιδέα το πώς θα δώσουμε πιο κρίσιμο και περίοπτο ρόλο στους ε, κοινωνικούς εταίρους στο επόμενο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε συμφωνούμε με το σχετικό εδάφιο της γνωμοδότησής σας ε, και το έχουμε σκεφτεί και από μόνοι μας στο σημείο αυτό. Τώρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα συνδέονται και με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων. Και η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα δραστήριες στην προώθηση και την εφαρμογή των βασικών αρχών του Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα αυτά. Και βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο ό,τι αφορά την υιοθέτηση νομικώς δεσμευτικών διατάξεων για τα θέματα αυτά. Έχαμε πρόσφατα ένα που οργάνωσε ο ΙΕ στη Γενέβη για το θέμα αυτό και εκεί ήταν ομόφωνη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη-μέλη ότι θεωρούμε κάπως πρόωρο αυτή τη στιγμή να υιοθετήσουμε ένα νομικά δεσμευτικό μέσο γιατί θεωρούμε ότι αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κατευθυντήριων δεν είναι αρκετό και θα πρέπει να το, να το επεξεργαστούμε περαιτέρω και χρειαζόμαστε μια συνένεση μεταξύ των ενδιαφερομένων. Αυτή η συνένεση είναι το ζητούμενο, γι' αυτό και θα την επιδιώξουμε. Οπότε η δέσμευσή μας για το μέλλον είναι να προωθήσουμε περαιτέρω τη, τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών και όχι τόσο σε αυτή τη φάση υπέρ ενός δεσμευτικά, νομικός δεσμευτικά, ε, δεσμευτικού μηχανισμού. Πάντως, όπως σας είπα, συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον ε, εισηγητή τον κύριο Παντζέρη, με την Εγκρίση Επιτροπή και με την Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Η κυρία Άλπιο Γκούσμαν φαίνεται να είναι στην ίδια γραμμή με την συλλογιστική της έκθεσης όταν λέμε για δεσμευτικές κοινωνικές ρήτρε. Και ο κύριο Γκέρεν, νομίζω έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση όταν είπε για τη Συμφωνία οικονομική εταιρική σχέση. Η αναπτυξιακή διάσταση πολύ αργά μπαίνει συνήθω στι διαπραγματεύσει ω στοιχείο και το αποτέλεσμα είναι σαφέ για μας που ασχολούμαστε με την ανάπτυξη. δεν είναι σοβαρή η αντιμετώπιση της εκρίζωσης της φτώχειας, της επισητιστικής ε, επάρκειας και ούτω καθεξής. Αν δεν κάνει την κατάσταση στο Μαλί καταλαβαίνει ότι η χώρα ήταν πολύ ευάλωτη. Πριν από λίγα χρόνια το Μαλί ήταν μια από τις ικανότερες αφρικανικές χώρες και ξαφνικά μετά τα όσα έγιναν στη Λιβύη ε, ε, έπεσε θύμα άνευ προηγουμένων ε, καταστάσεων με την εισαγωγή βαρέων πυροβολικών όπλων από την Λιβύη και σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κάποιο είδου παρατηρητήριο για τις ε, αρχικές ε, φάσεις ακόμα και για τα στάδια προτού προκύψουν οι σειράξεις. Επιμένω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε τις διάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπορεί να είναι δείκτης μια σύραξης που επίκειται. Δεν είμαι ακριβώς βέβαιο ότι μιλάμε για δύο πράγμα. Γιατί όταν λέτε για την εφαρμογή του πλαισίου ράγκη, πρέπει να συνεχιστεί και έχουμε αναλάβει δεσμεύσει, αλλά προφανώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη υλοποιεί κάποια στοιχεία αυτά για από, από αυτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τα ορυκτά των ε, συγκρούσεων. Δεν ξέρω λοιπόν τον, κατά πόσον είναι αντιφατικό να προβλέψουμε δεσμευτικού κανόνε και να είναι αντιφατικό με το πλαίσιο Ράγκη αφού οι κανόνε για τι επιχειρήσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει ούτω ή άλλω να εφαρμοστούν διεθνώ. Μπορούμε να έχουμε πολλά συγκεκριμένα νομικώ δεσμευτικά ε, εργαλεία για τη σχέση των επιχειρήσεων με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι ένα μόνο το μέσο. Ο κ. Ράγκη όταν ήρθε στο κοινοβούλιο πριν από λίγε εβδομάδε, κάτι ανάλογο μα είπε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 15 Δεκεμβρίου στι 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση 21 Ιανουαρίου. Για του συναδέλφου που ήταν εδώ από την αρχή, είπαμε ότι πρωτού ήρθε ο Επίτροπο έχουμε περίπου 20 λεπτά. Οπότε θα δούμε την έκθεση του κυρίου Νόιζερ για την ε, λευτική συμφωνία με τη Σενεγάλη, σημείο 11. Και αν προλάβουμε, θα ψηφίσουμε και αυτό το θέμα πριν τις 4.30. Οπότε να δώσω το λόγο στον κύριο Νόιζερ. Οι αλλιευτικές αυτές συμφωνίες είναι συμφωνίες για τις οποίες μόνο η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου χρειάζεται. Η Επιτροπή μας όμως καλό να τα συζητάει αυτά, διότι οι αλληλευτικές συμφωνίες έχουν μεγάλη σχέση με την ε, αναπτυξιακή πολιτική και στο παρελθόν είχαμε αρκετές διαφωνίες σε σχέση με επικείμενες ελληνικές συμφωνίες. Σήμερα λοιπόν θα δούμε την συμφωνία αυτού του είδους με τη Δημοκρατία της Ενεγάλης. Οι κανόνες σημαίνουν, ε, ε, ορίζουν ότι ναι ή όχι απλώς θα πούμε, χωρίς τροπολογίες, οπότε κύριε Νόιζερ έχετε το λόγο. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ ακόμα και αν είναι περιορισμένε οι δυνατότητες επιρροή που έχουμε, έχει σημασία η Επιτροπή ανάπτυξη να ασχολείται με αυτό το θέμα και με τι συμφωνίε τη αυτές τις αλληλευτικές, όπως και λόγω με τη Δημοκρατία της Ενεγάλης. Έχει σημασία να δούμε το νέο κανονισμό για την κοινή αλληλευτική πολιτική που θα πρέπει να προσαρμοστεί με τις συμφωνίες αυτές, γιατί μιλάμε για την αβιώσιμη αλληλεία και ε, είναι πολύ μεγάλη σημασία. Το είπατε κι εσείς, Πρόεδρε, και για μας, να ε, συντονιστούμε αυτά. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο δεν περιλαμβάνει την αλία σας που είναι το ψάρι του φτωχού είναι ευπρόσδεκτο αυτό. Αυτό ο αληφτικό φόρο υφίσταται υπερεκμετάλλευση από το Μαρόκο, τη Μαυριτανία, τη Σενεγάλη και τη Γουινέα Μπισάου και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέχει στήριξη μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη για την πρόθεση τη περιφερειακή διαχείριση τη φρύσα, δίνοντα προτεραιότητα σε όσου αλλιεύουν με τον πιο βιώσιμο τρόπο και συμβάλλουν στην επιστημιστική ασφάλεια και είναι ο πληθυσμό εκεί. Όσον αφορά την πρόσβαση στο Μερλούκιο, ε, που είναι ένας αλληλευτικός πόρος με κατάσταση αποθεμάτων αβέβαιη και υφίσταται επίσης υπερεκμετάλλευση, πρέπει να ακολουθεί η προληπτική προσέγγιση, η αρχή της προφύλαξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε στενά τις δραστηριότητες των μηχανοτρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τον τοπικό τομέα αλίας. Είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη των οποίων τα σκάφη αλλιεύουν στο πλαίσιο του πρωτοκόλου ανταποκρίνονται στις απαιτήσει για την υποβολή ετησίων εκθέσεων. Η χρηστή διακυβέρνηση προϋποθέτει τη διασφάλιση της διαφάνειας και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων καθ' όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλου. Αυτό θα μπορούσε να διευκολυνθεί μέσω τη κοινοποίηση των εκθέσεων τη Μικτή Επιτροπή Ελευτική Σύμπραξη στον τομέα τη Βέσμη Αλία και με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των ελευτικών κοινοτήτων, στις εργασίες τη μικτή επιτροπή. Χαιρετίζουμε ρητά τη στήριξη ύψους 750.000 ευρώ ετησίω για την ανάπτυξη του ελευτικού τομέα τη Σενεγάλης. Η ελόγω στήριξη ανταποκρίνεται στι ανάγκε τη δημοκρατία τη Σενεγάλης όσον αφορά την προώθηση τη επιστημονική έρευνα, τον έλεγχο και την καταπολέμηση τη παράνομη αλεία, καθώ και τη στήριξη τη αλεία μικρή κλίμακα, συμπεριλαμβανομένη αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, με σκοπό την αποκατάσταση των αποθεμάτων των ηχθιδίων. Υπό την έννοια αυτή νομίζω είναι σκόπιμο ως Επιτροπή Ανάπτυξης να συμφωνήσουμε και να καλέσουμε την Επιτροπή Αλίας ως αρμόδια επί της ουσίας να προτείνει στο Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του για την πρόταση απόφαση του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνία ελευτική σύμπραξη στον τομέα τη βιώσιμη αλεία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία τη Σενεγάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Νόρμπερτ. Δεν βλέπω κανένα συνάδελφο. Α, βλέπω ο κύριος Πόγκα θέλει το λόγο και μετά η Χάιντι Χάουταλα και άλλοι και ο κύριος Γκέρντς. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Νόισερ και τον υποστηρίζω στο θέμα αυτό. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κυρώσει τη συμφωνία αυτή στο βαθμό που υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση αλίας στη Σενεγάλη. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Πολύ σύντομος και μεστός και μπράβο σας. Ευχαριστώ η Χάιντι Χάουτ, αλλά και μετά ο Σολ Ευχαριστώ. Όντως, πολύ καλή αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση που συνοδεύει την πρόταση. Έχω όμως μία ερώτηση. Πώς θα ελέγξουμε την παράνομη, αδήλωτη και άναρχη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, έχει στενή συνεργασία με την Ιντερπολ και τα Ηνωμένα Έθνη για το θέμα της ε, παράνομης άναρξης και δήλωτης ελίας, γιατί είναι κέριο ζήτημα για τα αλληλευτικά αποθέματα. Δεν ξέρω αν είστε κατατοπισμένοι σχετικά ή μπορεί να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι ο συνάδελφος που έπρεπε να έρθει δεν, δεν πρόφτει. Α, συγγνώμη, έχει έρθει ο ο κύριος Πρέντα νομίζω ε, κατάφερε και ήρθε τελικά, δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχόλιο. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα της αλίας. Έχουμε επιτέλους νέες διατάξεις στην κοινή ελευτική πολιτική για να συνάπτουμε και καλύτερες συμφωνίες ελευτικής σύμπραξης. Ο Σαλ Γκέρενς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μου πείτε ο εισηγητής μας, είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι γίνεται σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση της συμφωνίας. Γιατί στο παρελθόν γινόταν ανάκληση αδειών, αλληλευτικών αδειών των, ε, ε των εταιριών που αλλίευαν ανοιχτά των αφρικανικών ακτών. Τι γίνεται, μήπως είναι απλώς ευσεβής πόθος να αποφευθούν τέτοιες παραβιάσεις. Αλλά τι συμβαίνει όταν πραγματικά διαπιστώνονται παραβιάσεις. Καλώ. έγιναν ερωτήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιο από την Γενική Διεύθυνση Μάρε, παρακαλώ, πείτε μας κι εσείς ποιος είστε και ετοιμάστε οι υπόλοιποι τις ε, κάρτες ψηφοφορίας γιατί θα ψηφίσουμε πριν έρθει ο Επίτροπος. Δίκλαος, ε, δεν ξέρω πώς προφέρετε ακριβώς το όνομά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Dominique Kleins και ερχάζομαι στο αρμόδιο τμήμα για τις διμερείς αλληλευτικές συμφωνίες στην Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έχω αναλάβει τη νέα συμφωνία και το αντίστοιχο πρωτόκολλο με τη Σενεγάλη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί αναγνώρισε τα πλεονεκτήματα της νέας συμφωνίας ε, και του πρωτοκόλου που προτείνουν οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, στηριζόμαστε στις αρχές της βιωσιμότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης, της συνέπειας και της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και φυσικά στηριζόμαστε και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Ο κύριος Νόιζερ περιέγραψε με σαφήνεια τις αδρές γραμμές της Αλληλευτικής Συμφωνίας και του πρωτοκόλου και εγώ θα απαντήσω απλώς στην ερώτηση για την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή πέραν στο, πέραν το, στο στο πλαίσιο της προτινόμενης συμφωνίας θα έχουμε κάποιες δράσεις για να βοηθήσουμε τους εταίρους μας να καταπολεμήσουν την παράνομη αδήλωτη και αναρχιαλία, IUU, και να σας επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει αναλάβει τη δέσμευση απέναντι στην κοινότητα δυτικοαφρικανικών χωρών και την κοινότητα κέντρο αφρικανικών χωρών να αναλάβει κάποιες δράσεις προκειμένου να αυξήσει την ασφάλεια της ναυτιλίας και της ναυσιπλοείας στον κόλπο της Γουινέας. Και οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ε, ένα σκέλος που αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Επίσης ε, εκπονούμε και σχέδιο δράσης που θα αφορά την περίοδο 2015-2020 και που θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της κατάστασης ασφάλειας στον κόλπο της ε, Γουινέας, την καταπολέμηση της πειρατείας, την πάταξη της παράνομης αλίας και οποιασδήποτε μορφής λαθρεμπορίου. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Um, you want to... Ευχαριστώ. Ο εισηγητής, δεν ξέρω Σάρλ, έμεινε ικανοποιημένο από τις απαντήσεις. Εγώ ρώτησα αν ε, επιβλήθηκαν κυρώσεις ή αν διαπιστώθηκαν παραβιάσεις που ε, προκάλεσαν την επιβολή κυρώσεων και αν ναι, τι είδους κυρώσεις επιβλήθηκαν και από ποιον. Δεν ξέρω, αν δεν έχετε πρόχειρη απάντηση μπορείτε να στείλετε και γραπτός ε, την απάντησή σας είτε προς εμένα, τη γραμματεία ή τον κύριο Γκέρνς. Βεβαίως, ε, εννοείται ότι για τις συμφωνίες της νέας γενιάς, τις νέες αλληλευτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανόμενε και αυτές που θέλουμε να συνάψουμε με τη Σενεγάλη, η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών αποτελούν καινοτομία. Σε ό,τι αφορά τέτοιες συμφωνίες και πρωτόκολλα, μέχρι στιγμής δεν είχαμε, δεν χρειάστηκε να λάβουμε μέτρα μετά από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ως κύρωση κυρίως την αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλου. Δεν προβλέπουν άλλη το κύρωση ή κάποια πιο στοχοθετημένη παρέμβαση κατά εφοπλιστών ή κατά εταιριών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια τη συμφωνία αυτή. Μάλιστα, αυτά για τις ελληνικέ συμφωνίε της Νέα Γενιά. Σάρλα, έχει να προσθέσει κάτι? Ομολογώ ότι δεν έμεινα ικανοποιημένο από την απάντηση. Βέβαια δεν φταίτε εσείς. Αλλά διαπιστώνουμε εδώ μια σημαντική έλλειψη σε ό,τι αφορά την επιβολή των κυρώσεων. Είναι σαν να έχουμε μαχαίρι, χωρίς ακορισμένη λεπίδα και χωρίς καν χερούλι. Είπατε ότι δεν ε, επιβλήθησαν κυρώσεις, που σημαίνει είτε ότι δεν έχουμε μηχανισμό ελέγχου, είτε έχουμε μηχανισμό ελέγχου που άκρος αναποτελεσματικό. Αυτή την έλλειψη θα πρέπει να την διορθώσουμε. Κατεπηγόντως, γιατί μέχρι στιγμής δεν επιβλήσαν ποτέ κυρώσεις, τι να πω. Μένω άναυδος. και συμφωνώ με την έκκλησή σας να μας ταλεί γραπτή απάντηση για τους ελέγχους. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Έγιναν έλεγχοι, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις και αν ναι, επιβλήθηκαν κυρώσεις. Παρακαλώ γραπτό στην απάντηση. Ναι, έχουμε μια νέα γενιά συμφωνιών που εφαρμόζονται από τώρα, αλλά τι έγινε στο παρελθόν σε περίπτωση που διαπιστώθηκε παραβίαση, επιβλήθησαν κυρώσεις και ο νέος κανονισμός με τι νέες διατάξεις προσπαθεί να καλύψει το, ίσως το προηγούμενο κενό. Μήπως θα μπορούσατε λοιπόν να στείλετε γραπτή απάντηση στον κύριο Γκέρνς, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να ψηφίσουμε, γιατί μα περιμένει και ο Επίτροπο. Θα ψηφίσουμε για να δούμε το αποτέλεσμα. Έχουμε μία πρόταση, μία τροπολογία του κύριου Γκέρνης, μία ψηφοφορία μόνο, άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody voted? Ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας. 17. Η απαρτία, ή όλοι όσοι ήταν εδώ, ε, ψήφισαν υπέρ. Εγκρίνεται η έκθεσή σας κύριε Νόιζερ. Και κύριε Πρέντα, θα ξανάρθουμε στα θέματα ελευθερικών συμπονιών στο μέλλον. Ο Επίτροπος είναι εδώ, θα περάσουμε πολύ γρήγορα στην ε, ομιλία του Επιτρόπου. Όσοι πρόκειται να φύγετε, παρακαλώ ησύχως. Just say, να θυμίσω ότι υπάρχει μια συνεδρίαση των σχεδόν για τα ορυκτά των συγκρούσεων που θα γινόταν εδώ στις 6.30. Η πρότασή μας είναι πλέον να γίνει αμέσως αφού ολοκληρώσουμε. Περίπου στις 5.45. Συνεδρίαση λοιπόν της ε, συνάντηση της ομάδας των σκιωδών αμέσως μετά την τη λήψη της συνεδρίασης. Παρακαλώ όσοι είστε στην ομάδα αυτή να μείνετε εδώ μετά. Και όσους θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους από τη γραμματεία το προσωπικό για να ξέρουν πότε θα γυρίσουν. Um, Συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον Επίτροπο για την Διεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη, τον Εύαν Μίμητσα. Ε, μόλις εδώ και ένα μήνα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του και είναι πάρα πολλά τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε. Μόλις μου είπε ότι χθε αργά επέστρεψε από τη Γουινέα, από το Κονάκρι, ε, στη Δυτική Αφρική και ξέρουμε ότι εργάζεται σκληρά από τη στιγμή που ανέλαβε. Και παρόλα αυτά θα ακούσουμε με μεγάλη χαρά τι ε, σκέψει για το Ευρωπαϊκό Έτο Ανάπτυξη. Επιτροπέ, ήταν ε, πολύ καλή στιγμή να έρθετε τώρα. Έχουμε και όλη τη συζήτηση για το θεματολόγιο για μετά το 2015. Το θέμα για το κλίμα είναι πάρα πολλές προτεραιότητές μας και θέλουμε να δούμε κατά πόσον μπορούμε να πετύχουμε μαζί επιτυχία αποτελέσματα. Θέλουμε λοιπόν τη σκέψη σα το πρόγραμμα και τι περιμένετε από το πρόγραμμα της Επιτροπής που θα μας αποκαλύψετε την ερχόμενη εβδομάδα επισήμω στο Στρασβούργο. Τόσα άλλα επίσης που έχουμε να πούμε. Έχετε τον λόγο, Επίτροπε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή Λίντα, αξιότιμη ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε συνεδρίες της Επιτροπής Ανάπτυξης ε, από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου πριν από ένα περίπου μήνα. Οπότε θα ήθελα καταρχάς να διατρανώσω τη σταθερή μου και στεναρή δέσμευση για στενή συνεργασία και συνεχή διάλογο μαζί σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι κέριο εταίρο σε σημαντικά θέματα στη διαδικασία μετά το 2015 και επίση στη συζήτηση για το πλαίσιο μετά το Κοτονού. Η για τα μακροπρόθεσμα διδάγματα που θα αντλήσουμε από την κρίση του έμπορα. Επίσης το Κοινοβούλιο θα είναι κύριος εταίρος για συγκεκριμένα θέματα που πολύ συχνά και τα επιμέρους θέματα είναι εξίσου σημαντικά με τη γενική στρατηγική. Γι' αυτό και είμαι θερμός υποστηρικτής ενός αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου σε, όλες, σε όλους τους τομείς που χρηματοδοτούμε, είτε με το Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας, είτε με το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ΕΤΑ. Θα επισέλθουμε σε λεπτομέρειες για τον κοινοβουλευτικό ρόλο αργότερα στη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με μία σαφή δέσμευση. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μερικές σημαντικές προτεραιότητες ε, που είναι αυτές που εντόπισα μετά από τον πρώτο μήνα άσκηση των καθεκόντων μου και μετά από συναντήσεις με ε, εταίρους στην Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το πλαίσιο των αηφόρων αναπτυξιακών στόχων μετά το 2015. Είναι αναμφίβολο ότι πιο εντυπωσιακέ πρόοδοι και πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά του αναπτυξιακού στόχου ε, αφορούν τομεί ε, των υφισταμένων αναπτυξιακών στόχων τη χιλιετία. Έχουμε όμω και πολλέ εκκρεμότητε. Το 2015 δεν θα είναι ένα καταληκτικό σημείο. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε του αναπτυξιακού στόχου τη ε, χιλιετία και να του αναπτύξουμε περαιτέρω. Την περασμένη εβδομάδα ο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων παρουσίασε την συνοπτική του έκθεση για το θεματολόγιο μετά το 2015, που θα συμβάλλει τα μάλα στι επικείμενε διακυβερνητικέ διαπραγματεύσεις. Επίσης, ε, ε, παρουσιάζει τα πορίσματα της ανοιχτής ομάδας εργασίας ως βάση για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Και τα έξι βασικά σημεία που επισημαίνει στην έκθεση του Γενικός Γραμματέας συνάδουν σε μεγάλο βαθμό και με τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δίνουν έμφαση στην αξιοπρέπεια, υπενθυμίζουν ότι η εξάλληψη της φτώχειας θα πρέπει να είναι ο γενικός ε, στόχος της βιώσιμης αναπτυξιακής ατζέντα και επίση τονίζει την ανάγκη της καταπολέμησης των ανισοτήτων. Επισημαίνει την έλλειψη αποκλεισμών ως σημαντική προϋπόθεση για κοινή ευημερία και επιβεβαιώνει ότι η δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ειρηνικέ κοινωνίε αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τη αηφόρου ανάπτυξη. Θεωρώ ότι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα στο ΙΕ συμπληρώνει την πιο διεξοδική και αναλυτική παρουσίαση της έκθεσης της Ανοιχτής Ομάδας Εργασίας και της ε, βιώσιμης αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Θα αποτελέσουν τη βάση για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την επόμενη 15 ετία και ε, αργότερα προκειμένου να εξαλειφθεί η φτώχεια, να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο και να προστατεύσουμε τον πλανήτη. Για να στεφτούμε επιτυχία οι βιώσιμοι στόχοι της ε, ε, ανάπτυξης ε, δεν αρκεί να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς. Το πιο σημαντικό είναι η ουσία, δηλαδή ότι η παγκόσμια κοινότητα θα επιδείξει τη βούληση και θα μεριμνήσει να εξασφαλίσει τα μέσα εφαρμογής και έναν αποτελεσματικό και αξιόπιστο μηχανισμό ε, παρακολούθησης για την αναθεώρηση της διαδικασίας. Επίσης θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά όλα τα μέσα εφαρμογής κάτι που προϋποθέτει μια ευρεία οικουμενική προσπάθεια μέσω της παγκόσμιας εταιρική σχέσης ε, για την αναπτυξιακή συνεργασία. Κάθε χώρα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να κάνει κτήμα ε, και να αναλάβει προσωπική ευθύνη για την ανάπτυξη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στις γενικές προσπάθειες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Οι κοινέ προσπάθειες με άλλους δωρητές, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Βραζιλία, θα αποτελέσουν ε, σημαντικό παράγοντα. Μία νέα και ενισχυμένη παγκόσμια εταιρική σχέση δεν θα πρέπει να αποκλεί κανένα και θα πρέπει να κινητοποιεί σε όλα τα επίπεδα τους ενδιαφερομένους σε όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, επιστημονικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινοβούλια και τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και αρχές. Ταυτόχρονα πιστεύω ακράδαντα ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας και πρωταθλήτρια στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε αυτή την ευθύνη θα πρέπει να την επομιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Θα πρέπει να εκπονήσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση με τα κράτη-μέλη και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να βαρύνουμε στη συζήτηση για τη ε, διατράνωση σημαντικών κοινών και φιλόδοξων στόχων και να ενθαρρύνουμε και τους επόλοιπους εταίρους μας να αναλάβουν ε, τις χρηματοοικονομικές και μη δεσμεύσεις τους ανάλογα. Πιστεύω ότι από κοινού θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση συνένεσης και στην σημαντική και θετική έκβαση ε, στην ε, τρίτη ε, διάσκεψη για τη χρηματοδότηση ανάπτυξης στην Αντίσα τον επόμενο Ιούλιο και στην διάσκεψη κορυφής το Σεπτέμβριο και το μετά το 2015 και στη διάσκεψη των Παρισίων για το κλίμα. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία υπερψήφισε το ψήφισμα για την κατάσταση μετά το 2015, έκθεση Steer για τους αναπτυξιακούς στόχους. Με το μήνυμα αυτό στέλνεται ένα χειρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και ενισχύεται τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μόλις επέστρεψα από το Ιγουινέα και θα ήθελα να αναφερθώ στην επιδημία του έμπολα. Η σοβούσα επιδημία του έμπολα είναι μια τραγωδία για τις χώρες και τους λαούς που χρήζουν της αποφασιστικής μας υποστήριξης. Όπως ξέρετε, ο συνάδελφος Χρήστος Τηλιανίδης συντονίζει τις κοινέ μας προσπάθειες για την καταπολέμηση της άμεσης κρίσης. Μέχρι στιγμής καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ένα πακέτο αντίδρασης ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα στηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο τις χώρες αυτές μετά το πέρας της οξίας κρίσης ή μετά την θέση της υποέλεγχο. Η αναπτυξιακή μας συνεργασία θα έχει κρίσιμο ρόλο κέριο ρόλο στην υπέρβαση των νέων και παλιών διαρθρωτικών προβλημάτων των χωρών αυτών. Η κρίση του έμπολα βάζει σε δοκιμασία και τον οικονομικό τομέα, αλλά και την οικονομία και τη διακυβέρνηση στι χώρε αυτέ. Και στι συζητήσει μου με τον πρόεδρο της Γουινέα και τον πρωθυπουργό, σχολείες αυτές τις προκλήσεις και μετά από μία επίσκεψη και σε τοπικό νοσοκομείο διαπίστωσε πόσο σημαντικό είναι να παράσχουμε στοιχειώδη ατροφαρμακευτική περίθαλψη στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η στρατηγική μας αναπτυξιακή επικεντρώνεται στη Γουινέα, τη Λιβυρία και τη Σιέρα Λεόνα και έχει διτό χαρακτήρα. Καταρχήν θέλουμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο της κρίσης ε, στις οικονομίες και τις κοινωνίες των χωρών αυτών και απ' την άλλη θέλουμε να αποκαταστήσουμε και να εξοπλίσουμε υγιείς ε, δομές σε τοπικό επίπεδο, να αναβαθμίσουμε οι υγειονομικές ε, συνθήκες και να βοηθήσουμε στην εξασφάλιση και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Μάλιστα έχουμε ένα περιφερειακό πρόγραμμα 28 εκατομμυρίων προκειμένου να βοηθήσουμε τις χώρες που έχουν πληγεί από το έμπολα στα πλαίσια των αναπτυξιακών προσπαθειών που αφορούν την αποκατάσταση και την παροχή ανακούφισης. Τα κονδύλια αυτά θα είναι πολύ χρήσιμα και θα τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερομένων χωρών από τον Ιανουάριο. Μάλιστα πρόσφατα, χθες, ανήγγειλε ένα νέο αναπτυξιακό πακέτο ύψους 62 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων συνεπειών της έμπολα στις τρεις χώρες. Το μισό από το, το πακέτο αυτό αφορά την Γουινέα. Οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα οικονομικά προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες δημοσιονομικής υποστήριξης και να, εξετάσουμε, να ε, ετοιμάσουμε νέες συμβάσεις δημιουργίας θεσμών. Πάνω από 148 εκατομμύρια ευρώ έχουν κινητοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λάβουν τη μορφή δημοσιονομικής υποστήριξης για την πρόθεση των ικανοτήτων των κυβερνήσεων για παροχή κοινοφελών υπηρεσιών και διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη νέα περίοδο, την ενδέκατη περίοδο του ΙΔΕΦ, e για να στηρίξουμε την διαδικασία ανάκαμψης σε καθοριστικού τομείς όπως την εκπαίδευση και τη γεωργία. Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Λιβερία, την Σχέρα Λεώνα και την Γουινέα έχουν ολοκληρωθεί. Ε, στον προγραμματισμό τους. Πρέπει όμως να έχουμε και ειδικά προγράμματα για την ε, λειτουργία των σχολείων όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ένα άλλο σημαντικό τμήμα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας για την ε, καταπολέμηση του έμπολα είναι η έρευνα. Για αυτό το σκοπό η έρευνα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του έμπολα θα πρικοδοτηθεί με άλλα 280 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Horizon 2020 για να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας στην ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων και να σώσουμε περισσότερες ζωές ανά τον κόσμο. Η τιμή των εμβολίων και ε, η κάλυψη του κόστους για τον εμβολιασμό κατά του έμπολα θα είναι ένα από τα ζητήματα του θεματολογίου μας και των προτεραιοτήτων μας για την αναπτυξιακή στήριξη στο υγειονομικό ε, σύστημα των ε, διαφόρων συνεργαζόμενων χωρών. Μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο Αντιπρόεδρο Μογκερίνη, τον Επίτροπο Ανδρουκάητη και τον ε, Συντονιστή Επίτροπο για τα θέματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του έμπολα, τον κ. Στυλιανίδη, θα έχουμε μία διάσκεψη ψηλού επίπεδου για τη μακροπρόθεσμη απόκρισή μα στον έμπολα στι αρχέ του 2015. Κυρίε και κύριοι, του χρόνου θα αρχίσουμε να μελετούμε και έναν ανανεωμένο πλαίσιο για τη συνεργασία μα με τι χώρε ΑΚΕ και την Αφρική. Η Συμφωνία Κοτονού είναι η πλέον συνολική συμφωνία Βορρά και Νότου στον κόσμο. Ε, σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος έχουν αλλάξει καθοριστικά από την ε, σύναψή της τον Ιούνιο του 2000. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους ΑΚΕ για να δούμε πώς θα μπορέσουμε περισσότερο να βελτιώσουμε την εταιρική μας σχέση στο μέλλον ώστε να έχει τα, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να βασιστεί τα αποτελέσματα της διαδικασίας για το διάστημα μετά το 2015 και να αντικατοπτρίζει τη διαφορετική κατάσταση των διαφόρων χωρών ΑΚΕ. Ε, καλωσορίζω το γεγονό ότι η ομάδα των χωρών ΑΚΕ ήδη μελετά πώς θα πρέπει να προχωρήσει. Η σύνοδος ΑΚΕ που έχει θεσπίσει μια ομάδα εξεχουσών προσωπικότητων το Δεκέμβριο του 2012 υπό την προεδρία του ε, Ομπασάντζο, του πρώην Προέδρου της Νιγηρίας. Εκεί συμμετέχουν 12 ε, εξέχουσες προσωπικότητες των χωρών ΑΚΕ με ένα ιστορικό ε, διεθνούς πρωταγωνιστικού ρόλου. Έχουν αναλάβει να μελετήσουν το μέλλον των σχέσεων των χωρών ΑΚΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η έκθεσή του θα υποβληθεί στην επόμενη Σύνοδο ΑΚΕ, τη οποία ημερομηνία θα οριστεί σύντομα. Μαζί με την Ένωση, μια ευρεία διαβούλευση και διάλογο για την διαδικασία μετά την Κοτονού θα ξεκινήσει κάπου του χρόνου. Ε, αναμένω την ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ίσως η Επιτροπή, σας θα μπορούσε να ορίσει έναν μόνιμο εισηγητή για τη διαδικασία για το διάστημα την Κοτονού, αλλά βεβαίως αυτή είναι μια απόφαση που θα λάβει το Κοινοβούλιο. Τώρα, ως προς τις θεματικές προτεραιότητες, σε αυτή τη φάση θα ήθελα να αναφέρω τουλάχιστον δύο ζητήματα που κατά την δική μου την άποψη πρέπει να τύχουν τις τη προσοχή μας και των ενδιαφέροντός μα. Τις ανισότητες και τα θέματα των φύλων. Οι ανισότητες είναι μια σοβαρή τροχοπέδη στην βιώσιμη ανάπτυξη ανά τον κόσμο. Οι ανισότητες ως προς την πρόσβαση στο νερό, στα τρόφιμα, το υγειονομικό σύστημα, την εκπαίδευση ή την υγειονομική περίθαλψη ε, και την υγιεινή. Ε, όλες αυτές οι ανισότητε στα δικαιώματα τη γη και τη μικροπιστώση ή τα δημοκρατικά, τις και πολιτικέ διαδικασίε και άλλα πολλά που θα μπορούσα να αναφέρω είναι σημαντικά και σε πολλέ περιπτώσει παίρνουν μεγαλύτερε διαστάσει. Αυτή είναι μια σοβαρή απειλή για οποιαδήποτε διεθνή, περιφερειακή ή διμερή προσπάθεια συνεργασία ανάπτυξη. Είμαι αποφασισμένο να δώσω αγώνα κατά των ανισοτήτων και να το θέσω αυτό το θέμα στο κέντρο των πολιτικών μου προσπαθειών. Οι ανισότητε συχνά σχετίζονται και με το φύλλο. Η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών είναι μέρο των εκκρεμουσών υποθέσεων μεταξύ των στόχων ανάπτυξη τη χιλιετία που προανέφερα. Δεν υπάρχει περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση φτώχεια να περάσει στο παρελθόν εάν δεν γίνουν σοβαρές και ταχείες βελτιώσεις στη ζωή των γυναικών και κοριτσιών σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είμαι λοιπόν αποφασισμένος να εξαλείψω και να καταπολεμήσω κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Πρέπει να υποστηριχθεί η συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις τομείς δράσης. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική σφαίρα επίσης. Το ε, υπάρχον πρόγραμμα δράσης για την ισότητα των φύλων εκπνέει του χρόνου. Φιλοδοξία μου είναι να αντικατασταθεί από ένα ανανεωμένο, ενισχυμένο θεματολόγιο ε, με συγκεκριμένου στόχου για να προωθηθεί η ισότητα των φύλων. Κυρίε και κύριοι, σε λιγότερο από ένα μήνα το Ευρωπαϊκό Έτο για την Ανάπτυξη 2015 πρόκειται να ε, ξεκινήσει. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να δείξουμε στου Ευρωπαίου, ιδίω στου νέου Ευρωπαίου, πόσο σημαντική είναι η αναπτυξιακή μα συνεργασία. Να του δείξουμε πώ οι εταίροι μα ανά τον κόσμο μπορούν να υποφεληθούν από τη στήριξή μα. Για να δείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί και η ίδια να ωφεληθεί από τη συνεργασία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα φιλοδοξότατο πρόγραμμα. Έχουμε ήδη ε, μία ιδέα για το πώς θα πρέπει να γίνει η οπτική μας προβολή, ένα κοτή εργαλείων για την ενημερωτική εκστρατεία και άλλο υλικό που θα μπορούσε να διαθέσουμε στους εταίρους μας. Υπάρχει ένα, ένας ειδικός ιστότοπος σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδεικνύει το πόσο σκληρά έχουμε εργαστεί στον τομέα της ανάπτυξης και για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έμφαση σε συγκεκριμένες ιστορίες και με 12 θεματικούς μήνες για την εκπαίδευση, τις γυναίκες και τα κορίτσια, την βιώσιμη ανάπτυξη ανάπτυξη μέχρι τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα που θα απασχολήσουν την εκστρατεία μα καθ' όλη τη διάρκεια του έτου. Είναι πολύ καλό που το Κοινοβούλιο με ενθουσιώδη τρόπο συμμετέχει, συνεστηρίζει τι προσπάθειέ μα, οργανώνοντα εκδηλώσει, ε, συμβάλλοντα τι ε, Ευρωπαϊκέ ημέρε ανάπτυξη, την ΕΞΠΟ, τη Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου, οργανώνοντα δημόσιε συζητήσει και επίση συμπεριλαμβάνοντα τα εθνικά κοινοβούλια. Κυρίε και κύριοι, ε, ε, κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα να ε, καλύψω και άλλα θέματα σε αυτή μου την εισήγηση, όπως την πολιτική συνοχή, ε, αλλά δεν υπάρχει αρκετός χρόνο, σε κάθε περίπτωση όμως για όλα αυτά, να μένω την συνεργασία του Κοινοβουλίου για να έχουμε μια φιλόδοξη αναπτυξιακή πολιτική στην Ευρώπη τα ερχόμενα χρόνια και τις δεκαετίες που επικίνδυνται, με τη στήριξη του ευρωπαϊκού κοινού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Με πολύ χαρά άκουσα πολλά από όσα είπατε. Για το θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε την ημερομηνία και δεν θα συμπίπτει με την Ολομέλεια στο Στρασβούργο γιατί ήταν δύσκολη αυτή η προηγούμενη κατάσταση. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε την εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη. Έχουν ζητήσει το λόγο ήδη αρκετοί συνάδελφοι με τη σειρά. Ο κύριος Πρέντα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εξ ονόματος της ομάδας του. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ και για τα όσα είπατε. Απευθύνομαι σε σας πάνω απ' όλα ως μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών και φυσικά εκτίμησα, όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, τη δέσμευσή σας και ε, τις υποσχέσεις ε, που δώσατε κατά τη διάρκεια ε, της ακρόασής σας. Και θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε, το αναφέρατε στο τέλος τώρα της παρέμβασής σας, θα θέλαμε, λέω, να μάθουμε και να γνωρίζουμε πώς εξελίσσονται αυτές οι δεσμεύσεις που αναλάβατε. Τι συνέχεια έχει δοθεί από την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων σας και μετά. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με την εξής ιδέα. Η έκθεσή μας για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία δεν θα μπορούσε να συνοδεύεται ε, από μία ανακοίνωση για να έχετε πιο πολιτικές προτάσεις για να βελτιωθεί η ε, υφιστάμενη πρακτική. Πώς το βλέπετε αυτό. Εκτός από την έκθεση και πέρα από την έκθεση να έχουμε και μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να θίξουμε και αυτό το πιο πολιτικό σκέλος, την πιο πολιτική αυτή διάσταση. Δεύτερον, ε, πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτή την πολιτική στο θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015. Και επίσης μιλήσατε για τη συνεργασία σας με την κυρία Μογκερίνη, αλλά ε, έχετε ε, ανταλλάξει απόψεις με την κυρία Μογκερίνη για να συντονίσετε την πολιτική αυτή. Μιλάμε πάντα για συντονισμό της αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά χρειάζεται και συνεργασία και συνεννόηση και συντονισμός των δικών σας υπηρεσιών με την κυρία Μογκερίνη, που είναι και την πρόεδρος κατά τα άλλα και είπατε πρόσωπος. Γιατί καλός είναι ο ευρωπαϊκός συντονισμός, αλλά θα πρέπει και οι εταίροι μας, κυρίως στα πλαίσια του ΩΣΑ να συντονίζονται. Αυτά. Και πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά που σας βλέπουμε. Καλά, για φέτος μπορεί να είναι, αλλά γενικότερα σας ξαναδούμε του χρόνου. Καλά, μέχρι τα τέλη του έτους δεν νομίζω να έχουμε άλλη συνεδρίαση. Ε, ο κύριος Πρέντα είναι συντονιστής της συνοχής. Ε, για την ανάπτυξη, όπως είπα. Ο κύριος Νόιζερ και μετά ο κύριος Γκέρανς. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ από πλευρά μου, πρώτα απ' όλα για το γεγονός ότι ήρθατε αμέσως ε, στην αρχή της θητείας σας και μάλιστα και πήγατε αμέσως και στις περιοχές που πλήττονται από τον έμπολα. Αυτό είναι ένα σαφές ε, σημάδι αλληλεγγύης και δεν δείξατε μόνο αλληλεγγύη αλλά δεσμευτήκατε και για οικονομικές υποσχέσεις. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω που χρησιμοποίησατε την πρώτη ευκαιρία πριν από λίγε μέρες στο Στρασβούργο να έρθετε στην συνάντηση ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ε, έκανε εντύπωση όχι μόνο σε εμά, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους συναδέλφους από τις χώρες ΑΚΕ. Πραγματικά ε, και μου το είπαν και οι ίδιοι. Αρχίσατε λοιπόν με ένα πολύ μεγάλο συν την θητεία σας και αναφέρατε και τις βασικές σας προτεραιότητες και μεταξύ αυτών τη Συμφωνία Κοτονού και τι θα γίνει την περίοδο μετά το 2020. Και κάνατε και μια ενδιαφέρουσα πρόταση που νομίζω θα πρέπει να τη συζητήσει η Επιτροπή μας να διοριστεί να οριστεί ένας μόνιμος εισηγητής για την ε, περίοδο μετά το Κοτονού. Και σε σχέση με την κρίση του έμπολα θα ήθελα να ξαναρωτήσω, όπως και ο συνάδελφος Πρέντα, πώς συντονίζεστε με την κυρία Μογκερίνη, αλλά και τον κύριο Στυλιανίδη, που και ο ίδιος μετέβη και στις χώρες που επλήγησαν ή πλήττονται από τον έμπολα. Κάνετε συνεννοήσεις μεταξύ σας, συμφωνείτε πώς θα γίνει επιμερισμός εργασίας και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μια παρουσία εκεί. Και επίσης να θυμίσω και κάτι. Η κρίση του εμπόλα μας έδειξε και πάλι πόση σημασία έχει διαρθρωμένη συνεργασία ε, στα πλαίσια της υγείας και στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε χώρες που είναι ακόμα ασταθείς. Ε, με τέτοιες επιδημίες ε, θα πρέπει με την πρόληψη και τη σωστή ιατρική, την προληπτική ιατρική να τις προλάβουμε. Όπως έδειξε και το παράδειγμα των γειτονικών χωρών, οι οποίες εμφάνισαν κρούσματα, τα οποία ελέγχθησαν όμως πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συστήματα υγείας ε, αυτών των χωρών, πώς να μπορέσει να τα ενισχύσει στο μέλλον για να υπάρξει καθολική υπηρεσία παροχής υγειονομικών υπηρεσιών υπήρξε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2010, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παγκόσμια Υγεία ονομάζεται αυτή η πρωτοβουλία και το πρόγραμμα δράσης και καλό θα ήταν να το συμπεριλάβετε και στο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Σαρλ Γκέρντς και μετά η Μαρίνα αλμπια Γκουσμάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ανακαλύψαμε έναν επίτροπο πάρα πολύ αποφασισμένο ενθουσιασμένο επίσης ε, σας ευχαριστώ να διατηρήσετε αυτή την ε, όρεξη και την ε, διάθεση που έχετε. Αξίζετε όλη μας τη συμπάθεια, αλλά ξίζετε και τη συμπόνια μας. Διότι στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, έχετε εταίρους. Για να το πω πιο συγκεκριμένα, έχετε και πεθερές που έχει και λόγο υπεθερά στον προγραμματισμό. Έχετε αδέλφια ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναν αδελφό που ασχολείται με το κλίμα και θέλει να σας πάρει τα λεφτά, <laughs> για να το πω έτσι με πάρα πολύ ομό τρόπο. Έχετε μια αδελφή που ασχολείται με το εμπόριο και ε, ε, έχετε και συγκρούσεις με όλους αυτούς τους συγγενείς στο περιβάλλον σας, πεθερές και αδέλφια. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει ενωμένης από τον ίδιο τον Επίτροπο, αλλά και τους υπαλλήλους που κάθονται εδώ εξεβονίμων, ε, διατηρεί πάντα την ευγένειά της σε όλες τις περιστάσεις. Εμείς καμιά φορά μπορούμε και τα λέμε πιο έξω από τα δόντια. Και πρώτος εγώ. Επανειλημμένα σήμερα το έκανα, ε, κάνοντας ερωτήσεις που με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, αν θέλαμε να εξηγήσουμε την ανάπτυξη σε αδαείς, και να εκδώσουμε ένα τέτοιο εγχειρίδιο για ασχέτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πηγαίνει προς την κατεύθυνση του 0,7% για την ανάπτυξη. Δεν θα το έχουμε καταφέρει το 2015. Είμαστε ο να αναδορητής, βασίζουμε την πολιτική μας σε κάποιες αρχές και σε κάποιες δράσεις. Αλλά μπορούμε να το δούμε και διαφορετικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσατε για ε, το στρατηγικό ε, πρίσμα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε το συντονισμό καλύτερα. Είπα ότι έχετε μια πεθερά και αδέλφια, ε, αλλά έχετε και εταίρους που είναι τα 28 κράτη-μέλη που κάνουν ε, το καθένα ακριβώς ό,τι θέλει. Και είδαμε στη διαχείριση του έμπολα τι εικόνα έδωσαν στην κοινή γνώμη με τη διαχείρισή τους. Επίσης έχω μεγάλη συμπόνια για τον συνάδελφό σας ε, που ασχολείται με την ανθρωπιστική βοήθεια, ε, που είναι ο κύριος Ηλιανίδης, με προκάτοχο την κυρία ε, Γεωργίεβα. Έρχεται λοιπόν το Συμβούλιο και λέει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους επιτρόπους, ότι ορίστε, έχετε κάποιον που θα είναι συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έμπολα. Θαυμάσια. Μπορεί να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χρειάζεται να του υπαγορεύει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του σώματος πώς θα ε, οργανώνεται εσωτερικά. Ε, μπορεί και η ίδια να διαβάσει τη συνθήκη για να κάνει το συντονισμό. Και μάλιστα είναι υποχρεωμένη να το κάνει αυτό. Να συντονίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης. Τα λέει ρητά η συνθήκη και επίμονα. Και θα ήθελα κι εσείς ως Επίτροπος να έχετε και το ίδιο κύρος. Ε, τουλάχιστον εμείς σας υποστηρίξουμε όσο μπορούμε. Πέρα λοιπόν από αυτό το μικρό εγχειρίδιο που θα εξηγεί ε, την ανάπτυξη χρειάζεται συνοχή και συντονισμός. Τα αναφέρατε και εσείς ο ίδιος. Και επιμείνατε στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα που θα βρείτε μπροστά σας ε, την επόμενη πενταετία. Έτσι λοιπόν είστε εσείς ο στρατηγικός μας εταίρος όλα αυτά τα θέματα. Και θα σας παρακαλούσα και εσάς και εμάς να σκεφτούμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ξέρω ότι όταν κάνουμε απευθεία άμεσε ερωτήσει, δεν έχουμε πάντα τις απαντήσεις. Χρειάζεται ένα πλαίσιο ε, να γράφονται όλα αυτά για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και σε σχέση με την προηγούμενη θητεία, Στι ζώνες των συγκρούσεων χρειάζονται κάποιες διαιτησίες να γίνουν για την ε, αρμπιτράζ, ε, για τη συνοχή και συνεκτικότητα των πολιτικών. Αυτό ποιος το αποφασίζει. Ε, θα μου πείτε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν διυπηρεσιακές ε, συσκέψεις. Δεν μου αρκεί αυτό. Όταν υπάρχουν συγκρούσεις σε βάθος θα πρέπει εσείς να έχετε το απαραίτητο κύρος ε, για να αποφασίσετε να βγάλετε μια απόφαση με τη δική σας κρίση και με ατράνταχτα στοιχεία. Εκεί χρειάζεται μια στρατηγική συνεργασία που εμείς επιθυμούμε και εσείς είμαι βέβαιος ότι συμμερίζεστε μαζί μας. Περιορίζουμε σε αυτά τα ολίγα σχόλια, ε, δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι η αποφασιστικότητα και το πνεύμα με το οποίο αναλαμβάνετε τα καθήκοντά σας είναι ελπιδοφόρα για να ε, προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλμπιόλ και μετά η Μαρία Χόρμπουργκ για να κλείσουν οι συντονιστές. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Τράτω με τις ευκαιρίες ε, για να σας ε, θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Πρόσφατα, χάρη σε μία διαρροή, είδαμε κάποια απόρριτα μηνύματα που δείχνουν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να, για να υπογράψει Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με, με το Εκοδόρ. Και μάλιστα φαίνεται ότι απείλησε το Εκοδόρ η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με κατάργηση ε, ανθρωπιστικής, ε, αναπτυξιακής βοήθειας αν δεν δεχτεί την συμφωνία αυτή. Φαίνεται ότι χρησιμοποιεί την αναπτυξιακή συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκβιάσει εταίρους της προκειμένου να συνάψουν συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Ως αρμόδιος επίτροπος για την ανάπτυξη θα επιτρέψει τη συνέχιση αυτού του εκβιασμού θα επιτρέψετε η αναπτυξιακή ενίσχυση να γίνει μέσω άσκησης πίεσης ε, προς συγκεκριμένες χώρες ε, ε, προκειμένου να συνάψουν συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που θα αφήνουν την οικονομία τους ξέφραγο αμπέλι για τις πολυεθνικές. Η κυρία αλλά από Πράσινους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση και χαιρετίζουμε όλη την δέσμευση και τη στράτευσή σας για την καταπολέμηση των διαφόρων μορφών ανισοτήτων. Ευπρόσδεκτη δέσμευση και αξιέπαινη. Και επίσης για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και την πάταξη κάθε μορφής διάκρισης βάρος των γυναικών ή περιορισμού των δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών. Όπως είπατε, υπερψηφίσαμε το ψήφισμα για τη διαδικασία μετά το 2015. Ελπίζουμε το ψήφισμά μας να εμπνεύσει το Συμβούλιο και να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας για τα γενετήσια και αναπαραγωγικά δικαιώματα νεαρών κοριτσιών και γυναικών. Ελπίζουμε και η θέση του Συμβουλίου να αντανακλά τις δικές μας θέσεις, γιατί σε πολλές χώρες του κόσμου δεν υπάρχει αυτή η δεδηλωμένη δέσμευση υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και νεαρών κοριτσιών για τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα. Επίσης θα πρέπει να επιμείνουμε στην προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, έκθεση του Γενικού Γραμματέου των Ηνωμένων Εθνών, που δημοσιεύθηκε στις 4 Δεκεμβρίου. Θα μπορούσατε να μας δώσετε πιο αναλυτικές πληροφορίες τώρα που δημοσιεύθηκε η έκθεση και θα ξεκινήσουν οι διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις τι οποίες θα διαδραματίσουμε ελπίζω σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιε είναι οι μείζονε προκλήσει ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ε, έναρξη των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πορίσματα της ε, έκθεσης ανοιχτής ομάδας εργασίας του Γενικού Γραμματέως, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές εν ώψη της διάσκεψης, παγκόσμιας διάσκεψης της Αντισαμπέμπα για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Διαπίστωσα ότι ο Γενικός Γραμματέας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη τα, μέλη, ε, τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, ε, προσελκύοντας ταυτόχρονα και ιδιωτικές επενδύσεις. Ποιε είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ λοιπόν εν ώψη της ε, επικείμενης ε, διάσκεψη κορυφή τη Αντισαμπέμπα για τη χρηματοδότηση τη ανάπτυξη. Ωραία. Αυτό είναι ο πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο να απαντήσει και μετά έχουμε και άλλου 10 περίπου μιλητέ για το δεύτερο γύρο. Είναι πολύ σημαντικό ποια είναι τα βήματα μετά το 2015. Έχουμε το Συμβούλιο της Παρασκευής, περιμένουμε κάποια συμπεράσματα για το ποια θα είναι η πορεία και στο εγκυσμένο, αλλά και στο απότερο. Έπεσαν βροχηδόν οι ερωτησει 5 5-6 λεπτά για να προλάβουμε και δεύτερο γύρο κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για, την, ε, για το ενδιαφέρον σα, τι ερωτήσεις, τα σχόλιά σας. Τα περισσότερα έχουν να κάνουν με τον ε, συντονισμό μεταξύ των επιτρόπων, των διαφόρων πολιτικών, των ευρωπαϊκών πολιτικών και πώς να δουλέψουν πραγματικά για την ανάπτυξη με έναν τρόπο συνεκτικό. Η νέα Επιτροπή νομίζω ότι όντως ε, αυτό που πρώτο έχει ως προτεραιότητα είναι ο συντονισμός των πολιτικών μας με μια τέτοια μεθοδολογία που οι αντιπρόεδροι να συντονίζουν ομάδες ή οικογένειες, για να το πω έτσι, πολιτικούς τομείς αρμοδιοτήτων των επιτρόπων. Μια από τις ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές ε, διαδικασίες συντονισμού ξεκίνησε στα θέματα των εξωτερικών υποθέσεων με την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη και πέντε ή έξι ε, επιτρόπους που ασχολούνται με θέματα εξωτερικών υποθέσεων αλλά και άλλα, την ενέργεια, τη γεωργία και είχαμε τουλάχιστον τρεις-τέσσερις συναντήσεις σε ομάδα αλλά και πολλές διμερείς συνομιλίες. Συμφωνούμε στη βασική αρχή που την πολιτική συνοχή θα την έφερνε στο, ε, στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μας ε, ε, προσέγγισης. Λόγου χάρη την επόμενη Παρασκευή, αυτή την εβδομάδα δηλαδή, θα έχουμε ένα συμβούλιο και με τα κράτη-μέλη δηλαδή και εκεί θα υποβάλουμε αυτήν την νέα προσέγγιση με μια κοινή εξωτερική και εσωτερική οπτική γωνία για τη μεταναστευτική πολιτική ή για το συντονισμό ε, στις εξωτερικές δράσεις. Αυτά ήδη φαίνονται στη διασύνδεση των τριών πτυχών των εξωτερικών υποθέσεων. Εξωτερική πολιτική και θέματα ασφάλειας, ανθρωπιστικές ε, άμεσες αποκρίσεις, ε, κρίσεις όλων των ειδών της κρίσης και ανάπτυξη. Ανάπτυξη για τις μακροπρόθεσμες λύσεις. Τον στηρίξουμε όλα αυτά τα στοιχεία ε, σε δύο φάσεις είναι το είδος της πολιτικής συνοχής που θέλουμε. Και νομίζω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. για να έχουμε μια τέτοια συντονισμένη εξωτερική δράση και ε, πολιτική στις εξωτερικές μας σχέσεις. Όλα αυτά Όλα αυτά ε, μπορούν να επιτρέψουν μια ευρωστότερη αναπτυξιακή πολιτική και όχι να ε, τμημα, τμηματικά να προσεγγίζουμε τους διάφορους πολιτικούς τομείς με, χωρίς να αξιοποιούμε συγκεκριμένες ενισφορές από άλλες πολιτικές. Υπήρχαν και κάποια άλλα συγκεκριμένα σχόλια για το συντονισμό για τα θέματα του έμπολα και γιατί ενδεχομένως να χρειαζόμαστε έναν Ευρωπαίο συντονιστή. Αλλά να πω ότι η κρίση του έμπολα, η τραγωδία του έμπολα είναι μια κατάσταση άνευ προηγουμένου, με διαστάσεις άνευ προηγουμένου που απαιτεί και άνευ προηγουμένου απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τη διεθνή κοινότητα. Γι' αυτό το λόγο οι προσπάθειες ε, συντονισμού πέραν του θεσμικού ρόλου και των ε, δυνατοτήτων της Επιτροπής ο συντονιστικός ρόλος ο δικός μας είναι πολύ σημαντικός αλλά το ίδιο και κάθε διεθνούς οργανισμού ή των εταίρων μας στην κάθε περιοχή. Για τις άμεσα αποκρίσεις λοιπόν υπάρχει συντονισμός προκειμένου να εντοπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες και να μεταφραστούν οι τεράστιοι αριθμοί του 1 δις ή του 1,1 δις της Ευρωπαϊκής Δέσμευσης ε, και των κρατών μελών της για την αντιμετώπιση των συνεπειών του έμπολα για να μεταφραστούν όλα αυτά σε κλίνες νοσοκομείων, σε φαρμακευτική στήριξη, σε ιατρικό προσωπικό στις χώρες που έχουν πληγεί από τον έμπολα. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό τώρα. Τουλάχιστον μια ιατρική ομάδα από κάθε κατός μέλος και αναβάθμιση της συντονισμένης μας δράσης. Αναμένω στη συνεργασία, την συνεργασία λοιπόν με τον συντονιστή Στυλιανίδη ώστε να υπάρχει μια, μια μακροπρόθεσμη απόκριση στην προσπάθειές μας και στην παρέμβασή μας κατά του έμπολα. Ε, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο θέμα του ενδεχόμενου εκβιασμού ή πίεση που λέγεται ότι δεν ξέρω ακριβώς ποιος η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει ασκήσει στο Εκουαδόρ για την σύναψη εμπορικής συμφωνίας, αλλά αυτό που ξέρω οπωσδήποτε και τα εμπορικά είναι σίγουρα το βασικό θέμα εδώ παρόλο που έχουν όλα αυτά σχέση και με την αναδείξη πολιτική. Ξέρω ότι εφόσον βρίσκονται υπό διαπραγματεύσεις οι συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας πάντοτε την αναπτυξιακή βοήθεια, τον προγραμματισμό για την ανάπτυξη, για τα αναπτυξιακά προγράμματα που μπορεί να πάυσουν ή να ανασταλούν μέχρι να υπογραφούν συμφωνίες. Αυτό είναι κάτι που πάντοτε ε, προκύπτει. Όλα τα διεθνή ενδεικτικά μας προγράμματα αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί και ε, υπογραφεί ασχέτως όμως των συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας. Άρα, εάν έχετε αποδεκτικά στοιχεία για τέτοιου είδους ε, δράσεις, σε καμία περίπτωση αυτού δεν συνάδει με την πολιτική που θα ήθελα να προωθήσω και για τις σχέσεις οικονομικών συμφωνιών με την όλη πολιτική μας για την βοήθεια προς άλλες χώρες δικαιούχους. για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015. Ναι, όντως, δημοσιεύτηκε η συνθετική έκθεση και τώρα την ε, μελετούμε κατά αλλά η πρώτη μου ενθερμό αντίδραση, το ανέφερα και στην σύγχυση μου, ήταν ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο-τρία στοιχεία που θα καθορίσουν την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πρώτον, υπάρχει μια ομαδοποίηση των στόχων που από 17 μπορούν να ε, συγκεντρωθούν σε έξι τομείς προτεραιότητας. Αυτό το θέλησαν το θέλουν οι περισσότεροι από εμάς και από τα κάτι μέλη. Υπάρχουν ακόμα κάποια διλήμματα, ανησυχίες για το εάν μπορούμε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση για όλη την πρόταση και να ξαναδούμε όλους τους στόχους ή να πάμε προς την κατεύθυνση της ομαδοποίησης αυτών των στόχων που τώρα επιβεβαίωσε και ο Γενικός Γραμματέας το ΙΕ. Είπε ναι, ας τους ομαδοποιήσουμε τους στόχους Αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει και η δική μας η θέση και να ξέρουμε πώς θα τοποθετηθούμε στις διπλωματεύσεις του χρόνου. Μετά η, συνοπτική αυτή, η συνθετική αυτή έκθεση αναφέρεται σε σημαντικά ζητήματα που σχεδόν μόνο εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τα ε, προωθούμε όπως την προσέγγιση των αναπτυξιακών πολιτικών μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καλή διακυβέρνηση. Αυτά έχουν τονιστεί ως μέρος των έξι θεματικών ενωτήτων στόχων και των τομέων προτεραιότητας. Έτσι θα μπορούμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις πραγματικά να απευθύνουμε έκκληση για μια διεθνή προσέγγιση τέτοιου είδους προς τα ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή και την προσέγγιση της ανάπτυξης μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, δηλαδή τα εργαλεία για την υλοποίηση που είναι εξίσου σημαντικά να πω ότι Εάν δούμε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις θέσεις του Κοινοβουλίου ώστε το 0,7 και οι δεσμεύσει μας να αναβαθμιστούν. Η δική μου προσωπική άποψη, διότι δεν τα έχουμε συζητήσει ακόμα στην Επιτροπή, ούτε με τα κράτη-μέλη ούτε εδώ στο Κοινοβούλιο. Η δική μου όμως προσωπική άποψη θα ήταν ότι για τη συνολική αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας, για την συνολική αποτελεσματικότητα της υλοποίησης, δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Σε όλα τα επίπεδα να δούμε μεταξύ των κρατών μελών τη νέα κατανομή μπορεί να υπάρξει, των δεσμεύσεών τους για την αναπτυξική βοήθεια, και μπορούμε να αναζητήσουμε και το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο για να πληρώσουν όλοι τις δεσμεύσεις τους, αλλά αυτή είναι η προσέγγιση που θα έπρεπε να επικρατήσει. Και έτσι θα έχουμε και μέσα διαπραγματευτικής πίεσης για να ζητήσουμε και από άλλους δωρητές να ενεργήσουν και να αναλάβουν και αυτοί τη δίκαιη δέσμευσή τους όπως τους αναλογεί, είτε είναι χρηματοοικονομική είτε όχι. Ε, στις διαπραγματεύσεις, γιατί για την ώρα μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όχι, η Ιαπωνία όχι. Έχουν άλλους τρόπους αναπτυξιακής βοήθειας και όχι μόνο την επίσημη αναπτυξιακή. Ε, πρέπει λοιπόν τώρα να αναζητήσουμε συμμετοχή από όλους, από όλους τους εταίρους διεθνέ επίπεδο, ώστε η επίσημη βοήθεια να γίνει πιο συνεκτική, να γίνει ισχυρότερη και για να υπάρξουν και άλλοι τρόποι, άλλες μορφές υλοποίησης με καλύτερα αποτελέσματα και πιο ορατά. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Έχουμε εννέα ομιλητέ. Θα σα παρακαλέσω ένα δίλεπτο καθένα στο πολύ. Δεν είστε υποχρεωμένοι να τα εξαντλήσετε, αλλά τουλάχιστον έτσι θα έχουμε χρόνο για όλου. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο στην Επιτροπή. Όπως είπατε, Πρόεδρε, είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά του και θέλουμε να συνεργαστούμε στενά μαζί του σε αυτό το έργο του. Στην αρχή είπε ότι και τα 28 κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δεσμεύσει και τους τις θύμισε. Και ε, εμείς οφείλουμε να ε, τους κάνουμε να τα τηρήσουν όλα αυτά. Αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αναλάβει δεσμεύσει. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το εξή. Δεδομένου ότι πρόσφατα έχει γίνει μεγάλη πρόοδος ιδιαίτερα στην πολιτική ε, της διατροφής και του επισητισμού για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Βέβαια είναι ακόμα τεράστιο σκάνδαλο και με συγκλονίζει ότι πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε βράδυ κοιμούνται πεινασμένοι και άλλα 2 δισεκατομμύρια υποσυτίζονται και πεινάνε. Και κατά τη διάρκεια της Ιλλανδικής Προεδρίας ε, ε, κυριάρχησε ένα σχέδιο για τη διατροφή και τον επισητισμό και την ε, υλοποίηση αυτό, και αυτό δεσμεύει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη-μέλη για να επιτευχθεί προοδός μετρήσιμη και ποσοτική. Τώρα ερωτώ τον Επίτροπο. Έχει γίνει πρόοδος έκτοτε από τα συμπεράσματα αυτά που συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο. Και δεύτερο, γνωρίζει ότι ε, ε, μια ομάδα παρακολούθησης από 10 κράτη-μέλη περίπου ολοκληρώνει μια έκθεση. Τι καθεστώς έχει αυτή η έκθεση και τι πρόοδος έχει γίνει και εκεί. Και ένα τελευταίο. Τι υποστήριξη χρειάζεται ο Επίτροπος από εμά, τους βουλευτές. Πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Επίτροπε. Εμείς πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να έχουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τον πρώτο μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες που μας παραθέσετε είναι σωστές. Τουλάχιστον ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Και μία από τις πολιτικές ανησυχίες ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Γραμματέως ε, ε, φαίνονται ότι συμπίπτουν. Καλό αυτό, καλό σημάδι και συμφωνώ με το σχόλιο σας για τα μέσα εφαρμογής. Γιατί μπορεί να έχουμε γενναιόδορους και φιλόδοξους στόχους, αλλά δεν έχουμε κατάλληλα μέσα εφαρμογής, θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εκπονήσει για το τέλη Ιανουαρίου την ανακοίνωσή της. Το Κοινοβούλιο θα καταρτήσει την έκθεσή του και μάλιστα εγώ θα συντάξω την έκθεση αυτή στην Επιτροπή ΝΤΕΒΕ για τα μέσα χρηματοδότηση μετά το 2015. Και αυτό το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τι προϋποθέσεις έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι αξιόπιστη σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις χρηματοδότησης που ίδια αθέτησε τα τελευταία χρόνια και τι νέα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να κινητοποιηθούν σε συνδυασμό με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα μέσα για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική που θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο αντιπρόεδρος μας Παύλο Βάιρινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για την πρόοδο που έγινε στην ομαδοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Και επίσης χαιρετίζω την το συντονιστικό ρόλο που θα παίξει η πατεκπρόσωπος Μογκερίνη σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές πτυχές της ανάπτυξης. Αλλά χρειαζόμαστε και ένα γενικότερο συντονισμό. Όπως είπατε κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας και αναπτυξιακής πολιτικής. Και επίσης ε, ε, έχουμε ηγετική θέση στην εμπορική πολιτική. Ε, εμπόριο και βοήθεια συμβαδίζουν. Και στις διαπραγματεύσεις του γύρου της Δόχα, στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, βασικός στόχος είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και κυρίως των λιγότερων αναπτυσσομένων χωρών. Και σίγουρα στην αναπτυξιακή βοήθεια σημαντικό στοιχείο παίζει και, είναι και το εμπόριο. Υπάρχει άρρηκτος δεσμός και το θέμα του περιβάλλοντος είναι συναφές. Και δεν μιλούμε μόνο για καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά και την πρόσπιση της βιοπικιλότητας και την ε, οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίω. Χρειαζόμαστε και ένα, και ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό σύστημα της ανάπτυξης παγκοσμίω. Ελπίζω λοιπόν ε, υπό το συντονισμό της κυρίας ε, Μογκερίνη θα έχετε καλή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ όλων αυτών των πτυχών ώστε να επηρεάσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αποτελεσματικά την παγκόσμια ανάπτυξη και φυσικά την αηφόρο ε, ανάπτυξη από κάθε άποψη. Τι γνώμη έχετε λοιπόν για αυτό το γενικό και παγκόσμιο εσωτερισμό που απαιτείται. Uh, um, Ευχαριστώ Επίτροπε, είστε μέλος μιας νέας επιτροπής που συνήθως καλείται να δώσει νέα ζωή στις αναπτυξιακές εταιρικές σχέσεις και τα αναπτυξιακά προγράμματα, να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να αντιμετωπίσει, όπως είπατε, τις νέες και δυσκολότερες προκλήσεις που προκύπτουν στην αναπτυξιακή συνεργασία. Δηλαδή αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η εικόνα, η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα, από τα αποτελέσματα των ε, προγραμμάτων. Δεν νομίζω ότι κάποια στιγμή να έρθει η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο με μια απόλυτα ξεκάθαρα στρατηγική για το πώ να βελτιωθούν οι ε, σχέσει συνεργασία μεταξύ των διαφορών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και αν έπρεπε να υπάρχει κάποια είδου συγχώνευση μεταξύ κάποιων οργανισμών ή φορέων. Και κατά δεύτερον, μπορεί να ξέρατε ότι είμαι ε, ο υπεύθυνο ομάδα ελέγχου ε, τη Επιτροπή μα, τη ομάδα Α και τα έγγραφα που λαμβάνουμε είναι μη δημοσιοβομενά και απόρριτα. Η ομάδα ελέγχου όμως έχει θέμα με το χαρακτηρισμό των εγγράφων διότι ακριβώς στα συμπεράσματά μας συμπεριλαμβάνεται σχόλιο για τα απόρριτα αυτά έγγραφα που μας αποστέλει η Επιτροπή. Όμως το Κοινοβούλιο πρέπει να λογοδοτεί στους πολίτες και είμαστε υπεύθυνοι για την δημοκρατική αξιοπαστία και τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει ψήφισμα για κάποιο μέτρο εφόσον θεωρεί ότι η Επιτροπή έχει ενεργήσει πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται για εκείνη από τις βασικές νομοθετικές πράξεις. Εάν εγκρίνει τέτοιο ψήφισμα το Κοινοβούλιο, μπορεί να το κάνει μόνο δημοσίως. Σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο του ε, εφαρμοστικού μέτρου της Επιτροπής και η απόκριση του Κοινοβουλίου σε αυτό ε, αναπόφευκτα θα δημοσιοποιηθούν. Δεν θα μπορούσατε λοιπόν να μας ξεκαθαρίσετε πώς να διασφαλίσουμε ότι η εργασία κοινοβουλευτικού μας ελέγχου γίνεται με το διαφανέστερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο για τους πολίτες μας, ώστε να ξέρουν γιατί στο όνομά τους δεν, ε, ότι εκπληρούμε τα καθήκοντά μας χωρίς να ε, μειώνουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω τον Επίτροπο κάτι ε, για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές ε, σύραξη. Το Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί, ο εισηγητής εδώ, για τη νομοθεσία σχετικά με την εισαγωγή τέτοιων ορυκτών από εμπόλεμες περιοχές. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση ε, ότι θέλει να ρίξει φως δηλαδή στα συναδευτικά μέτρα. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν το συζητάει πουθενά το Κοινοβούλιο, αλλά είναι σημαντικό στοιχείο εκτός από την νομοθεσία για να ε, επηρεάσουμε τα πράγματα κάπως επιτόπου. Η νομοθεσία, ξέρετε, αφορά μόνο την εισαγωγή εδώ και ε, κάποια εργοστάσια όπου τίκονται αυτά τα μέταλλα ή κάποια δηληστήρια. Ε, μόνο η ανακοίνωση όμως έχει δυνατότητα να επηρεάσει τα πράγματα στις περιοχές της ίδιας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σκέφτεται αυτά τα συνοδευτικά μέτρα που υποθέτω ότι θα χρηματοδοτηθούν και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης που αυτό το καιρό προγραμματίζει τον προπολογισμό του. Θα μας δώσετε και ένα χρονικό ορίζοντα. Πότε θα έρθουν αυτά τα συνοδευτικά μέτρα και πότε θα τεθούν σε ισχύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σλάι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν υπάρχει κάτι πιο ευχάριστο από το να σας ακούω να λέτε ότι θα αντιμετωπίσετε τις ανισότητες, ε, όπως είπατε και μεταξύ των κρατών και εντός των κρατών, ως προς τις ανισότητες και την πρόσβαση στους πόρους, τις διάφορες διαστάσεις που κι εσείς θυμήσατε προηγουμένως, νερό, ε, μόρφωση, υγιεινή, ε, εισόδημα, υπάρχουν και άλλα θέματα που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και που μπορεί να είναι επιτακτικής ε, ακόμα και αν αυτό δεν φαίνεται και επειδή δείχνουν ότι η ρίζα του κακού έχει διαφορετική αίτια, δηλαδή το μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης. Η δική σας ευαισθησία σε αυτά τα θέματα θα στηριχθεί πλήρως και από μένα και από πολλούς άλλους συναδέλφους πιστεύω και σε αυτή την Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Διότι στην έκθεση που υπερψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία πριν από λίγες μέρες, όλες οι ομάδες συμφώνησαν ότι ο αγώνας κατά των ανισοτήτων πρέπει να είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες μαζί με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εκρίζωση της φτώχειας. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπατε, ε, είναι, σημαντικό, είναι σημαντικός ο ρόλος του θέματος αυτού στις μελλοντικές μεταπραγματεύσεις, αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε με πυγμή όταν πρέπει να μιλήσουμε με ενιαία φωνή και με δυνατή φωνή. Εκεί θα μπορούσε να συνεισφέρει, είπατε, εκπρόσωπος Μογκερίνη. Η αποφασιστικότητα λοιπόν εδώ είναι βίωνη. Ε, και ελπίζουμε ότι με την δική μας συμβολή θα πείσουμε και τις ε, πιο διστακτικές κυβερνήσεις για το θέμα αυτό αντιμετώπιση των ανησυχητήτων. Και η σχετική έκθεση λέει ότι κανένας στόχος δεν θα έχει επιτευχθεί εάν δεν επιτυγχάνεται για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν τους στόχους ε, για την περίοδο μετά το 2015 θα πρέπει να ε, δούμε και την πολιτική συνεκτικότητα για την ανάπτυξη. Όπω είπατε την Παρασκευή, το Συμβούλιο θα κοιτάξει και τα συμπεράσματα που θα επηρεάσουν τη μεταναστευτική μα πολιτική ή η ομαδα μα. Θέλει λοιπόν συνοχή στι μεταναστευτικέ πολιτικέ που θα πρέπει να συνάδουν όχι μόνο με τι αναπτυξιακέ μα πολιτικέ, αλλά και με την ανθρωπιστική βοήθεια λόγου χάρη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώ προτίθεστε να κινηθείτε για να υλοποιήσετε αυτά τα φιλόδοξα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ήδη προβλέπετε κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Okay, the last three speakers, Maria Heubuck, Enrique. Ευχαριστούμε. Yeah, Maria. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε, ε, Μιλήσατε και για τις εμπορικές συμφωνίες, αλλά στις εμπορικές συμφωνίες ε, δεν είναι μόνο η άμεση σύνδεση με την αναπτυξιακή πολιτική, έχουν και έμεσες επιπτώσεις. Ας πούμε, αυτή η συμφωνία TTIP για τις επενδύσεις και το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, τι επιπτώσεις θα έχει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γενικά, ε, στο παγκόσμιο εμπόριο, πώς θέλετε να ε, προστατεύσετε τις χώρες που πλήττονται ε, από την ε, εξαγωγή κάποιων ουσιών και κάποιων ορυκτών που πρέπει να πληρώνουν δασμούς. Παντού κάθε χώρα θα πρέπει να μπορεί να έχει επισητιστική κυριαρχία, άρα να είναι σε θέση να προστατεύει ε, ε, την οικονομία της. Είπατε ότι η Γεωργία είναι ένας ε, τομέας κλειδί, όχι μόνο στην οικοδόμηση μιας οικονομίας μιας χώρας, αλλά και στην καταπολέμηση της ένδυας. Και πολύ συγκεκριμένα να ρωτήσω, να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα και στο θέμα των ανισοτήτων. Έχουμε ακόμα στο Ουσπεκιστάν ε, ε, καταναγκαστική εργασία ε, στον τομέα του βάμβακος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει πρόθεση να καταπολεμήσει αυτή την κατάσταση, αλλά παραμένει η κατάσταση αναλύωτη και απαράλλακτη και τα δεινά των εργαζομένων ανδρών και γυναικών. Τι θα γίνει λοιπόν ε, με αυτό το θέμα του Ουσπεκιστάν για να σταματήσει πραγματικά αυτή η καταναγκαστική εργασία. Θα χρειαστούν ε, ε, ακόμα 186 εκατομμύρια να δώσουμε σε αυτή τη χώρα για τη γεωργία της όταν διατηρεί αυτό το σύστημα της καταναγκαστικής εργασίας στα, στις βαμβακοφυτίες. Και πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα τερματιστεί μια τέτοια πρακτική. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ερίκε Γκερέρο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ζητώ συγγνώμη που δεν άκουσα την αρχική σας παρέμβαση, αλλά γνωρίζετε ότι στο Κοινοβούλιο συχνά συμπίπτουν ε, ταυτόχρονα συνεδριάσεις και έχουμε και άλλα καθήκοντα. Ε, θέλω να γνωρίσω την άποψή σας για τα εξής δύο. Πρώτον, για το συντονισμό των δωρητών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη θητεία ενέκρινε μια, μια, ένα αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταθέσει ένα κανονισμό ακριβώς για αυτό το συντονισμό. Από τότε καμία είδηση δεν έλαβαμε σχετικά. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε κανένα σχέδιο, το έχετε στο πρόγραμμά σας, ε, το πρόγραμμα εργασίας, το έχετε υπόψη σας, για να υπάρξει καλύτερο συντονισμός και να έχουμε και οικονομίες και πιο αποτελεσματική βοήθεια. Δεύτερη ερώτηση. Το 2015 θα γίνουν πολλές διεθνείς ε, διασκέψεις και μεταξύ αυτών είναι η έγκριση αναθεώρηση, δεν ξέρω, του σχεδίου ε, ε, δράσης 2005-2015 για τη μείωση των κινδύνων από τις θεομηνίες. Ξέρετε ότι όλη αυτή η πρόληψη και η μείωση του κινδύνου ευνοεί την καλύτερη αντιμετώπιση των κρίσεων και τη δυνατότητα υφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Και σας ρωτώ, το έχετε σκεφτεί ήδη, υπάρχουν κάποια στοιχεία στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με αυτή την ε, διεθνή διάσκεψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα και εγώ μια-δυο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα για το στόχο του 0,7% εάν κάποιες χώρες δεν ε, το έχουν χρησιμοποιήσει. Μήπως πρέπει να αφήσουν άλλες χώρες να αναλάβουν περισσότερη πρωτοβουλία. Αυτό θα το δούμε στις συνομιλίες για μετά το 2015 και για το πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη. Εδώ χρειάζεται να γίνει κάποια πρόοδος και ακούσαμε το τι φρικαλαιότητες ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τη Δημοκρατία του Κονγκό και στη Συρία ξέρουμε επίσης τι γίνεται ταυτόχρονα. Συζητήσαμε τον προπολογισμό και την απαλλαγή του 2014 με τα διαρκή προβλήματα, τα δημοσιονομικά που γνωρίζουμε. Πώς την Επιτροπή θα μπορούσατε να πιέσετε λίγο για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, να βρούμε κονδύλια για τα προγράμματα πρώτης προτεραιότητας και μετά για τη συνολική μας ε, συνεκτικότητα στην πολιτική, για τη συνοχή και την Αφρική. Μετά την περσινή σύνοδο, τι ε, συνέχεια δίδεται, πώς συνδυάζεται η ανάπτυξη με θέματα καταπολέμησης τρομοκρατίας, τι πολιτική συνοχή μπορούμε να δούμε προς την Αφρική. Ακούσαμε και τι έγινε στην Μεκτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ίση εκπροσώπηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσαμε για φτώχεια, για νέου χωρί δουλειά, χωρί προοπτικέ, που πολύ εύκολα γίνονται υλικό εκμετάλλευση από μεστές και τρομοκράτες. Υπάρχει μια πολιτική ε, θεώρηση για αυτά τα θέματα, για μια στρατηγική παρέμβαση. Αυτές τις λίγες ερωτήσεις, Επίτροπε. Είναι ο πρώτος σας μήνας, οπότε αν δεν τις απαντήσετε όλες μαζί μπορείτε να ξανάρθετε σε ένα μήνα. Thank Σας ευχαριστώ. Όντως, πληθώρα ερωτήσεων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις περισσότερες. Αλλά το βασικό είναι να, να κρατήσουμε ζωντανό και συνεχή διάλογο μεταξύ μας. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε. Οπότε εκφύσεως ο πρώτος διάλογος είναι και πιο γενικός. Πιο αναλυτική συζήτηση θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και στο μέλλον για επιμέρους θέματα. Μπορούμε για παράδειγμα να έχουμε μία ειδική συνάντηση για το θέμα του παγκόσμιου συντονισμού ή του συντονισμού της ε, αναπτυξιακής βοήθειας που δίνουμε ε, και το συνδυασμό με το θέμα των ε, ορυκτών που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Αυτό θα το δούμε στον τακτικό διάλογο που θα έχει ε, η Επιτροπή, η Επίτροπη με τις αρμόδιες επιτροπές. Τώρα, για τα επιμέρους θέματα. Μας ενδιαφέρει η επιστηστική πολιτική και ο υποσυτισμός ε, είναι σημαντική προτεραιότητα. Ο περιορισμός του υποσυτισμού είναι σημαντική προτεραιότητα της αναπτυξιακής ε, βοήθειας που παρέχουμε σε πολλές χώρες. Πρόσφατα συμμετείχα στη Ρώμη, στη δεύτερη παγκόσμια διάσκεψη για τον επισητισμό. Και επ' ευκαιρία διατρανώσαμε τις ε, δεσμεύσεις μας να ξεπεράσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας για τον επισητισμό και να θέσουμε τη διατροφή και τον επισητισμό ως ύψητη προτεραιότητά μας στους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έχουμε και μειώθηκε σίγουρα η πείνα, ο λοιμός, από τα 1,2 εκατομμύρια στους 1,2 δις 800 εκατομμύρια. Αλλά και 800 εκατομμύρια άνθρωποι που πεινάνε είναι υπερβολικός αριθμός. Ακόμη και 100 νηστικά παιδιά, 100 πεινασμένα παιδιά είναι υπερβολικός αριθμός. Δεν υπάρχει αποδεκτός αριθμός πεινασμένων ανθρώπων. Οπότε και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων επισητισμού που λάβαμε. Και οι σχετικές εκθέσεις μοιράστηκαν το Νοέμβριο στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και είμαστε σε θέση τώρα να περάσουμε στις έμπρακτες συνεισφορές και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε ό,τι φορά τις προτεραιότητές μας για τον επιστησμό στα πλαίσια της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Τώρα, συντονισμός κοινοτικών θεσμικών οργάνων και κρατών μελών. Είναι τριπλός αυτός ο συντονισμός. Καταρχήν θέλουμε καλύτερο συντονισμό των ε, προγραμμάτων αρρωγής με συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Και εκεί έχουμε εντυπωσιακή πρόοδο. Και βελτιώνεται και ο συνολικός συντονισμός με τους δωρητές, αλλά ιδιαίτερα με τα κράτη-μέλη. 40 χώρες στις οποίες έχουμε κοινά προγράμματα υπάγονται στην κοινή διαδικασία προγραμματισμού στην οποία συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και αυτές οι 40 χώρες εταίροι. Και 20 από αυτά τα κοινά προγράμματα ε, έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε σίγουρα έχει βελτιωθεί ο συντονισμός μας με τα προγράμματα των μεμονωμένων κρατών μελών στις χώρες εταίρους. Τώρα, στην, στο πρόγραμμα για την αλλαγή, στο θεματολόγιο για την αλλαγή, επικεντρώσαμε τα προγράμματα αρρωγής στις ε, υπανάπτυκτες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, της πλέον χρήσης βοηθείας δηλαδή. Και ακολουθούμε επιλεκτική προσέγγιση των τομέων. Εντοπίζουμε μέσα αφήνεια τους τομείς σε συνεργασία φυσικά με τη χώρα αποδέκτη, τη χώρα εταίρο. Και εκεί λοιπόν ο συντονισμός έχει, έχει βελτιωθεί. Εκεί που θα πρέπει να βελτιωθούμε είναι στο παγκόσμιο συντονισμό των δωρητών. Με τους ε, μίζωνες δωρητές και τους αναδυόμενους δωρητές. Με τις Ηνωμένε Πολιτείε καλά τα πάμε στο συντονισμό. Και έχουμε απτά παραδείγματα όπου πραγματικά λειτουργεί ο συντονισμός μας. Και πολύ σύντομα θα φτάσουμε σε επίπεδο αμοιβαία παροχής κάποιων χρηματοδοτικών μηχανισμών προγραμμάτων που τα διαχειριζόμαστε είτε εμείς είτε χρηματοδοτούνται από τους οργανισμούς μας. Και ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται εκεί και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ως προς την Κίνα, και εκεί υπάρχει αισιοδοξία για βελτίωση του συντονισμού. Πριν από 10 μέρες ήμουνα στην Κίνα και συζήτησα το θέμα του συντονισμού με τους ομολόγους μας στην Κίνα. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα αναπτυξιακά μας προγράμματα και οι αναπτυξιακές μας πολιτικές διαφέρουν. Εμείς επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, στις κοινωνικές υποδομές, στη συνδρομή σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, τη γεωργία, την υγεία, προγράμματα που αφορούν την επιστηστική ασφάλεια. Ενώ η κινέζικη αναπτυξιακή βοήθεια επικεντρώνεται περισσότερο στις επενδύσεις ή σε σχέδια υποδομών. Πάντως, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο καλός συντονισμό δεν σημαίνει αμοιβαία ε, κριτική ε, των διαφόρων αναπτυξιακών μοντέλων, ούτε ανταγωνισμό των επιμέρους αναπτυξιακών μοντέλων. Το θέμα είναι να καταστήσουμε συμπληρωματικά αυτά τα αναπτυξιακά μοντέλα ή να αυξήσουμε την συμπληρωματικότητά τους και όχι να επικρίνουμε ένα στο αναπτυξιακό μοντέλο του άλλου. Και η Κίνα είναι πρόθυμη και στερνίζεται αυτή την ερμηνεία του συντονισμού. Και έχουμε και τριμερή συζήτηση με την Κίνα για τις αναπτυξιακές μας πολιτικές ε, στην Αφρική. Οπότε είναι σημαντικός ο παγκόσμιος συντονιστός των δωρητών, γενικό συντονισμό των δωρητών και αποτελεί και δική μας προτεραιότητα. Στο θέμα του ελέγχου τώρα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά ταμεία και κονδύλια. Θα επαναρχόμαστε τακτικά στο θέμα αυτό και στην Επιτροπή σας και γενικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως νομίζω ότι βρήκαμε καλή συμβαστική λύση. Θα μπορέσουμε χάρη σε αυτή να βελτιώσουμε το στρατηγικό μας διάλογο. Βέβαια για το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας τα πράγματα είναι σαφή ε, και ξέρουμε πώς λειτουργεί ο έλεγχος και σε θεσμικό και σε πρακτικό επίπεδο. Αλλά για το Αναπτυξιακό ταμεία Είμαι διαλεκτικός και φιλόδοξος ως προς τον διάλογο μεταξύ μας. Και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θέλω στο θέμα αυτό να αξιοποιηθεί πλήρως. Με βάση φυσικά τα θεσμικά όρια και τις θεσμικές ιδιαιτερότητες είμαι έτοιμος και πρόθυμος να έχουμε και νέο γύρο συζητήσεων για τα θέματα αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε τίποτα να χωρίσουμε εδώ. Δεν είναι επίμαχο το θέμα μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής ή μεταξύ Επιτροπής ΔΕΒΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ. Θέλουμε τη μέγιστη δυνατή ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο αυτό και στο στρατηγικό διάλογο. minerals, yes. Για τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως όντως και κατά τη διάρκεια της ακρόασής μου εδώ στην Επιτροπή σας. Πώς να το πω. Ε, έδειξα αλληλεγγύη θεσμική ε, όσο, εξ όσων θυμούμε, θα θυμάστε και εσείς, σας ζήτησα, ας αφήσουμε λίγο χρόνο, ένα-δύο χρόνια, να δούμε πώς αυτή η διαδικασία οικειοθελούς πιστοποίησης θα λειτουργήσει και ε, από κοινού να αξιολογήσουμε στη συνέχεια ε, αν θα χρειαστεί κάτι πιο δεσμευτικό ή υποχρεωτικό ως μέτρο για το εμπόριο για ε, τις ε, πόλεμες περιοχές και τα ορυκτά από εκεί. Ε, ε σέβομαι απολύτως το συλλογικό πνεύμα και τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το, το έχω συζητήσει και με βουλευτές και με επιτρόπους, συναδέλφους μου και πρέπει να πω ότι ίσως χρειαστεί να ξανακουβεντιάσουμε το πλαίσιο τους περιορισμούς που υπάρχουν, ε, το κόστος και το όφελος ε, μιας ενδεχόμενης ε, υποχρεωτικής διαδικασίας ή συστήματος ή νομοθεσίας με δεσμευτικό χαρακτήρα για τα ορυκτά από τις εμπόλεμες περιοχές. Γιατί εάν πάρουμε αυτό το δρόμο, δεν είναι απαραίτητο πάντα το νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να δίνονται και κίνητρα ενδεχομένω για τους ενδιαφερομένους να εμπλακούν. Σε συνεργασία όμως με τις υπηρεσίες ε, της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για το εμπόριο, είμαστε πρόθυμοι να τα κοιτάξουμε αυτά τα θέματα, ε, αλλά με ευρύτερο πνεύμα για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Είναι γνωστά, είναι δεδομένα τα προβλήματα σε αυτό το τομέα. Τι άλλο έχουμε. Μια στιγμή να δω. Ε, trade, ε, Λοιπόν, για το εμπόριο. Ε, μιλήσατε για την επιρροή των εμπορικών ζητημάτων ε, της αναπτυξιακής πολιτικής, δηλαδή πώς, πώς επηρεάζει ε, τις ε, χώρες με τις οποίες έχουμε αναπτυξιακές σχέσεις. Ποτέ εγώ δεν θεώρησα ότι το μόνο κίνητρο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι το εμπόριο ή του ιδιωτικού τομέα ή γενικότερα της οικονομίας των κρατών αυτών που είναι εταίροι μας. Πάντα ε, βλέπω το εμπόριο συνδεδεμένο και σε ε, συνάφεια με τα κίνητρα που δίνουμε και στον ιδιωτικό τομέα για να αναβαθμιστεί η δυνατότητα των χωρών αυτών και της διακυβέρνησης και της οικονομίας τους για να μπορέσουν να υποστηρίξουν ιδιαίτερα ε, πολύ μικρές αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες τους. Και μόνο αν έχουμε μια τέτοια οικονομική θεώρηση, με καλύτερα ανεπτυγμένο δυναμικό, μπορούμε να ανοίγουμε τις ευρωπαϊκές αγορές για το εμπόριο. Ιδιαίτερα στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, με τη διευκόλυνση του εμπορίου. Έτσι θα αναπτυχθεί και θα ανθίσει και ο ιδιωτικό τομέα και μόνο αυτή είναι η σωστή οδό κατά τη γνώμη μου για την ανάπτυξη και τα σωστά κίνητρα επαναλαμβάνω. Για τα θέματα της καταναγκαστικής εργασίας. Βεβαίως αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το γενικότερο θεματικό πρόγραμμα και τα προγράμματα που ε, εκπονούμε. Είτε πρόκειται για θέματα φύλου, για την παιδική εργασία. Ξέρετε, είναι μια σειρά ζητημάτων όλα αυτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες ε, τέρους μας. Πάντα θεωρούμε ότι η καταναγκαστική εργασία είναι προτεραιότητα για μας, η καταπολέμησή της. Υπάρχουν χώρες ε, με τις οποίες υπάρχουν ε, εθελούσεις διαδικασίες για τη μείωση ή την εξάλληψη τελείως της ε, καταναγκαστικής εργασίας. Σκέπτομαι εδώ την ε, ειδική πρωτοβουλία του 2015, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανάπτυξης και τα αναπτυξιακά προγράμματα να εστιαστούν περισσότερο σε αυτά τα θέματα. με συγκεκριμένες δράσεις δηλαδή για τη μείωση και πλήρη εξάλληψη της ακαταναγκαστικής εργασίας. Στη γεωργική παραγωγή αλλά και στη βιομηχανία σε σειρά κρατών. Για τη μείωση των θεομηνιών βεβαίως θα συμμετέχουμε πλήρως στην ε, διεθνή διάσκεψη στην Ιαπωνία, στο Σεντάι θα γίνει αυτό. Συνεισφέρουμε κι εμείς γενικότερα για τη μείωση του κινδύνου, για μια βιώσιμη ανάπτυξη και με βάση τους στόχους μας για να προλαμβάνουμε θεομηνίες. Βέβαια, μέχρι την επόμενη διάσκεψη δεν πρόκειται να υπάρξει ένα ε, πλαίσιο ολοκληρωμένο, αλλά σε ό,τι αφορά τις δικές μας δράσεις και την ε, συνεργασία μας για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά θα πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες δράσεις για να μειωθούν οι θεομηνίες και οι κίνδυνοι θεομηνιών και καταστροφών, είτε αυτές είναι φυσικές είτε είναι ανθρωπογενείς. Βέβαια, έχουμε περιορισμού στα δημοσιονομικά μας που επηρεάζουν ήδη από τώρα το αναπτυξιακά μας σχέδια, έργα και προγράμματα. Θα σας τα πει αυτά ο Γενικός Διευθυντής. Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς, στην επιλογή των πληρωμών που μπορούμε να κάνουμε για φέτος, έχουμε κάποιους περιορισμούς, τα γνωρίζετε, για την αναπτυξιακή μας συνεργασία. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να ε, χρηματοδοτούμε στο ακέραιο τα προγράμματα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Υπάρχουν και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών πάρα πολύ δραστήριες αλλά τα κριτήρια για την επιλογή και τη μείωση των πληρωμών είναι αρκετά ευαίσθητα και θα πρέπει για πρώτη φορά να μπούμε σε αυτή την ε, επίπονη διαδικασία κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και δυστυχώς και του χρόνου. Θέματα ασφαλείας και ανάπτυξης και πάλι είναι αλληλένδετα πάρα πολύ μεταξύ τους και δεν νοείται φυσικά ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια ή χωρίς ένα σταθερό πλαίσιο. Or, or in the ε, Είτε πρόκειται για μια συγκεκριμένη χώρα εταίρα μας, είτε για μια περιφέρεια. Αλλά δεν νοείται ασφάλεια από την άλλη και σταθερότητα, δεν υπάρχει μια αναπτυξιακή προοπτική σε μια χώρα. Ξέρετε, λοιπόν, αυτά είναι ένα διώνυμο. Πάνε χέρι-χέρι η ανάπτυξη και η ασφάλεια. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ε, υιοθετήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση της τρομοκρατίας ή της ασφάλειας σε κάποιες χώρες με τα αναπτυξιακά προγράμματα και μέσα. Αλλά καμιά φορά μας προβληματίζει ο τρόπος. Ε, θα χρειαστεί ίσως ένα νέο πολιτικό και νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσουν καλύτερα αυτά τα πράγματα. Γιατί τώρα έχουμε ακόμα κάποιες ανησυχίες, ερωτηματικά για το πώς θα χρηματοδοτηθεί ας πούμε μια δράση ε, στην ασφάλεια, μια επιχείρηση. Τι παίρνουμε ένα κονδύλι ε, και το μεταφέρουμε κάπου αλλού. Έτσι, ίσως θα πρέπει στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη να τα ξαναδούμε αυτά από κοινού. Να υπάρξει ας πούμε νέος νομικός τρόπος, πλαίσιο, χρηματοδοτικό, για να υπάρξει πλήρης ε, και αποτελεσματική διασύνδεση της ανάπτυξης με την ασφάλεια. Νομίζω ότι τα απάντησα όλα περίπου ή τα περισσότερα μη τι άλλο. Α, και η μετανάστευση. Ήταν ένα από τα θέματα που τέθηκαν, αλλά νομίζω ότι το κάλυψα προηγουμένως. εξωτερικός και εσωτερικός. Υπάρχουν στοιχεία και πτυχές που σύντομα θα περιληφθούν στις προτεραιότητές μας για τις προσεχείς εβδομάδες με τα κράτη-μέλη. Θα περάσουμε σε στενότερες συζητήσεις του ρόλου της ανάπτυξης για την πρόληψη ή την καταπολέμηση της λάθρου μετανάστευσης. Αυτό όμως θα είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Αυτό που χρειάζεται να δούμε είναι τι θα κάνουμε από κοινού με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής. Και θα φροντίσουμε να υπάρξει ε, συμπόρευση των δύο αυτών διαστάσεων της εξωτερικής και εσωτερικής αντιμετώπισης της μετανάστευσης με ένα πολύ ε, σαφές πακέτο μέτρων όπου θα φροντίσουμε να γίνει σαφές τι και πώς τι σημαίνει μετανάστευση και πώς μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές πτυχές της μετανάστευσης. Και εσωτερικός και εξωτερικός. για τις χώρες εταίρους, τις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Επίτροπε, απαντήσατε πάρα πάρα πολλές ερωτήσεις. Θέλετε να προσθέσετε κάτι πάρα πολύ γρήγορα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εδώ έγινε μια παρανόηση ε, θα ήθελα να μιλήσω για δεσμευτικά ή μη δεσμευτικά μέτρα βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι είστε αρμόδιος για να θέσω ένα τέτοιο θέμα. Εγώ ρώτησα για την επικοινωνία που είναι δική σας ε, ευθύνη και το κατά πόσον έχετε προβλέψει μέτρα για να γίνει η βιώσιμη εξόριξη ε, κάτι που να υλοποιείται, που να, να γίνει πραγματικότητα τι προβλέπετε να κάνετε, πώς θα το υλοποιήσετε, τι ε, χρηματοδότηση προβλέπετε από το ενδέκατο πλαίσιο για την ανάπτυξη και τι επικοινωνία υπάρχει. Δεν ανάγκη να μου τη δώσετε τώρα αυτή την απάντηση, γραπτός κάποια άλλη στιγμή, απλώς να το σκεφτούμε που έχουμε φτάσει. Κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα. Πρέπει να παραδεχτώ για το δεσμευτικό ή όχι των μέτρων δεν το έχουμε καλύψει ακόμα. για το τι θα γίνει με τα ορυκτά των ε, συγκρούσεων και το τι μέτρα θα λάβουμε τώρα για τα εμπορικά και τα αναπτυξιακά στοιχεία του ζητήματος. Θα τα δούμε. Νομίζω η καλύτερη δυνατή συνεισφορά της αναπτυξιακής ατζέντα μας και του Επιτρόπου της Ανάπτυξης θα είναι να υπάρξει κάποιο είδους επικοινωνία ή μία λεπτομερέστερη και προσεκτικότερη καταγραφή του τι συμβαίνει στις περιοχές παράνομης εξόρυξης και σε εμπόλεμη κατάσταση όπου υπάρχει εκμετάλλευση ορυκτών. Επίτροπε, ευχαριστούμε που ήρθατε απόψε. Μείνατε παραπάνω 20 λεπτά από το χρόνο σας. Ελπίζω να μην σας καθυστερήσαμε από κάτι. Ευχαριστούμε για τις απόψεις σας και αναμένουμε τη συνεργασία μαζί σας και στο μέλλον. Επειδή είχαμε κάνει τα προηγούμενα σημεία ήδη, έχουμε ολοκληρώσει για σήμερα, εκτός και αν δεν υπάρχει κάτι κατεπήγον, δεν έχω ειδοποιηθεί για κάτι τέτοιο, οπότε κηρύσω τη λήξη της συνεδρίασης και να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση εμάς είναι στις 21 Ιανουαρίου και 22. Είναι πολύ νωρί, έτσι μοιάζει, για να πει κανεί καλά Χριστούγεννα, γιατί θα βρεθούμε και την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Αλλά για όποιον δεν δω, ε, να περάσετε καλά στι γιορτέ και εσεί το ίδιο, κύριε Επίτροπε για το ε, νέο τόσο πρόκειται σε δύο εβδομάδες περίπου.